Πάντοτε περιμένει κανεί από του πολιτικού ε, ηθήνοντε να έχουν και μια δεύτερη επιλογή, μια δεύτερη εναλλακτική. Πείτε μα ποια είναι αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάλπελτ, για ένα λεπτό.